Ε, έλεγξε την ε, εντολή των ε, κυρίων των πρόβλης Σόζιεν, Αλεξάνδερ Γκάμπελιτ, Ζαν Κάρλο Σκοτά και Ντανίλο Όσκαρ Λαντσίνη και πρότεινε να, να επιβεβαιώσουμε την εντολή τους η οποία ξεκινά αντιστοίχω από 19 Μαρτίου, 4 Απριλίου, 17 Απριλίου και 17 Απριλίου του 2018. Υπάρχουν ενστάσει, η εντολή εγκρίνεται.